του ασφάλιστου, γιατί οι πολίτε στην παρούσα κρίση χάνουν την εμπιστοσύνη του για την Ένωση. Α φροντίσουμε εδώ τουλάχιστον να μην γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Έχουμε τώρα την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για την μη βιώσιμη αλληλεία σκουμπριού στο, βορειο, βορειοανατολικό Ατλαντικό. Καταρχάς, ο συντάκτης της ερώτηση έχει το λόγο για πέντε λεπτά, ο κύριος Γκάλαγκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να θέσω αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα για τη μη βιώσιμη αλληλεία σκουμπριού στο Ατλαντικό. Ατλαντικό. Μιλάμε ε, για ανεύθυνη, ε, ανεύθυνο καθορισμό ποσοστώσεων που έχουν θέσει η Νίση Φερόε και η Ισλανδία για το 2013. Ε, Μιλάμε για αύξηση από το 1% στο 23% και αυτό πραγματικά θα απειλήσει τη βιωσιμότητα των εχθεαποθεμάτων σκουμπρίου και την πελαγική αλία το Συμβούλιο, το Θαλασσίο ε, Συμβούλιο έχει σταματήσει, έχει ε, καταργήσει από μέλη της αυτές τις δύο ε, χώρες λόγω αυτών των πρακτικών τους, οι οποίες θα έχουν επιβλαβέστατη επίπτωση στην πελαϊκή αλία. Θα έπρεπε η υπεραλίευση και άλλων ειδών να μας είχε κάνει να καταλάβουμε ότι είναι επικίνδυνο, όπως με την περίπτωση του ψαριού προσφυγάκη λοιπόν της 100 το 2006 ήταν η ποσόστοση, αφαιρώ 23% φέτος. Από 4,6 ε, έχουν αυξήσει ε, σε περισσότερο από, 2000, ε, από 23% το 2012 και η Ισλανδία έχει επίσης ε, αυξήσει, έχει ξαπλασιάσει το μερίδιό της, 52% πλέον ε, υπερβαίνεται από αυτό το οποίο επιστημονικά θα ήταν βιώσιμο. Αυτές οι ανεύθυμενες αλληλευτικές πρακτικές είναι και αντίθετες και με την ε, νομοθεσία 1026 ε, και ακόμη χειρότερα οι νήσοι Φερόε έχουν φύγει και από τις διευθετήσεις των πέντε παράκτιων ε, χωρών και για τη ΡΕΚΑ Ατλαντικού Σκανδιναβία και λένε ότι θα αυξήσουν σημαντικά το μερίδιό του. Θα πρέπει η Κομισιόν, επειδή έχει εντολή ε, πολύ ισχυρή, δεν θα πρέπει να την παραγνωρίσει, θα πρέπει πλέον να δράσει ε, βασισμένη ακριβώ αυτή την πολύ ισχυρή εντολή που έχει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ω εισηγητή σα καλό πραγματικά να λάβετε άμεσα δράση. Έχει περάσει ε, ο καιρός για λόγια και πρέπει να δούμε πλέον έργα για να σώσουμε αυτή την βιομηχανία, αυτόν τον κλάδο. Υπάρχουν συγκεκριμένε απαιτήσει στο σχέδιο κανονισμού. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά για μένα να καταλάβω για ποιο λόγο η Κομισιόν και οι Επίτροπο συνεχίζουν να αγνοούν τι απόψει των περισσότερων βουλευτών του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να βλέπετε, πιστεύω, ότι η υπεραλίευση αυτή πραγματικά θα οδηγήσει σε καταστροφή ε, του κλάδου. Υπάρχουν τουλάχιστον 12 γύρια διαπραγματεύσεων όπου κανένας μάλλον μέρος δεν έδωσε σερλιστικές προτάσεις. Μόνο ε, αν λάβουμε άμεσα δράση θα έχουμε αποτελέσματα. Εγώ ε, κατηγορώ την Κομισιόν για όλη αυτή την κατάσταση. Ούτε πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ε, θα φροντίσουμε για τη βιώσιμη αλίευση του Σκομπρίου αν δεν επιβάλλει και τις απαιτούμενες κυρώσεις η Κομισιόν. Η Ισλανδία, τα Φερόε αυξάνουν τα μεριδιά τους με τεράστιες ποσότητες. Πολύ σκληρά μέτρα εσωτερικά στην Ένωση έχει λάβει κομισιόν και τα υποστηρίζω. Κατά της Ισπανίας, για παράδειγμα. Αυτό μπορεί να ε, δείξει ε, ότι εμεί θέλουμε να υπάρχει βιώσιμη αλία. Ο πρόεδρος Επιτροπής Αλίας, Γκαμπριέλ Μάτο, μου ζήτησε να κάνω ε, αυτή τη ε, δήλωση, απουσία του, και λέω ότι και η και η νήσι Φερό δεν φέρονται ανεύθυνα. Θα πρέπει να αλλιεύουν βιώσιμα. Και αντί να μειώσουν κατά 15% με βάση επιστημονικές ε, συμβουλές ε, το μερίδιό τους, το αυξάνουν στο 23%. Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι η Κομισιόν ήταν στην πρώτη γραμμή και πάντοτε έλεγε ότι πρέπει να έχουμε βιώσιμα εχθεία αποθέματα και βιώσιμη αλία. Και όλοι το υποστηρίζουμε. Δεν βλέπουμε όμως αυτό να αντικατοπτρίζεται στις αποφάσεις που δεν λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχετε μέχρι τώρα αναλάβει δράση για την αποτελεσματική σωστή εφαρμογή μέτρων εμπορικών μέτρων για την αποτροπή αυτής της κατάφορης ανεύθυνης ε, αλληλευτικής πρακτική αυτών των δύο εταίρων. Τώρα πρέπει να δράσουμε και όχι αργότερα. Έχετε λάβει μια ισχυρή εντολή, αλλά την αγνοείτε κυρία Επίτροπε την εντολή του σώματο. Και εγώ πραγματικά χάνω την εμπιστοσύνη μου και ανησυχώ, ανησυχώ για το μέλλον, για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Ειλικρινά ελπίζω να έχετε να μα δώσετε απόψε κάποια καλά νέα, κάποιε καλέ ειδήσει και να μα πείτε ότι τώρα θα λάβετε υπόψη σα ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα λάβετε την δέωσα δράση. Ευχαριστώ. Η κυρία Δαμανάκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάλαχερ που έθεσε το θέμα. Σημαντικό θέμα όντως. Το συζητήσαμε και εδώ στο παρελθόν τις συνέπειες της υπεραλίευσης από την Ισλανδία και τα Φερόε στα αποθέματα αυτών των ειδών. Πρέπει να σας πω ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες του Κύριε Γκάλαχερ για τον αντίκτυπο που έχουν οι αυτέ του δικού δικούς μας ιδίω Ιδίως τον αντίκτυπο των δράσεων αυτών στις τοπικές αλληλευτικέ κοινότητες, στα μικρά σκάφη, τους μικρούς ψαράδες που δεν έχουν εναλλακτικέ. Συμφωνώ ότι για αυτού η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Παρακολουθούμε λοιπόν προσεκτικά την κατάσταση. και μέσω κάθε διάβλου προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση της Ισλανδίας, στην κυβέρνηση των νησιών Φερόε για να αλλάξουν την πολιτική τους. Ελπίζουμε ότι στο τέλος παρότι θα πάρουμε χρόνο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσει με όλες τις παράκτιες κυβερνήσεις και να υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία για τα αποθέματα. Δεν συμβαίνει βέβαια κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε λοιπόν. Συνοψίζοντας, η επιλογή των εμπορικών κυρώσεων είναι επιτάπητος. Συζητείτε. Είναι σημαντικό ωστόσο να εξετάσουμε προσεκτικά δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες. Πρώτον, τις νομικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούμε και δεύτερον, τη χρονική στιγμή των δράσεών μας. Για τους κουμπρί. Συζητούμε με τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή τις πιθανές εναλλακτικέ λύσεις. Την άλλη εβδομάδα θα συναντήσω τον οδηγό υπουργό της Βρυξέλλες και ελπίζω ότι θα υπάρξει κοινή απόφαση. Θέλουμε να υπάρξει κοινή απόφαση με την οδηγική κυβέρνηση για το θέμα. Να σας πω ωστόσο ότι η Επιτροπή ήδη εξέτασε τις ε, διαδικαστικές ε, διαστάσεις για να επιταχύνουμε τη διαδικασία λήψη αποφάσεως αν αποφασίσουμε να προχωρήσουμε. Αν αποφασίσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε ήδη έχουμε όλες τις ε, προετοιμασίες έτοιμες. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα σας ενημερώνουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό την επόμενη εβδομάδα όταν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με την οδηγική κυβέρνηση. Αυτά για το σκουμπρί. Τώρα, για τη ρέγκα του Ατλαντικού. Σαφέστερη δυστυχώς είναι εδώ η κατάσταση θα έλεγα. Προφανώς η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για την αγγελία που έγινε στις 26 Μαρτίου από πλευράς νησιών Φερόε που μονομερός υπερτριπλασίασαν την ποσόστοσή τους. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Επίσης, απαράδεκτο είναι ότι εγκατέλειψαν τις πολυμερείς συζητήσεις, την τράπεζα των πολυμερών διαπραγματεύσεων. Και η Επιτροπή και οι Νορβηγή εταίροι μας, με κοινή δήλωση, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας και ζητήσαμε από τα νησιά Φερόε να ανακρούσει πρίμνα αμέσως. τονίζοντας ότι αυτές οι μονομερείς, μονομερείς πράξεις επηρεάζουν σοβαρά την ε, βιωσιμότητα των αποθεμάτων. Όπως σας είπα, εδώ το τοπίο είναι σαφέστερο. Και έδωσα το πράσινο φως για να ξεκινήσει η εσωτερική κοινωτική διαδικασία, ε, διαδικασία της Επιτροπής για την χρήση των εμπορικών ε, μέσων κατά των νησιών Φερό. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η διαδικασία. Ευχαριστώ. Οι αγορητές των πολιτικών ομάδων τώρα για το ΕΛΚ. Κύριος Βαρέντσα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που συζητούμε το θέμα της αλίας στην Ισλανδία, γιατί κάποια στοιχεία μας, δεν μας έχουν ε, ικανοποιήσει. Αυτή μονομερή, ο μονομερής καθορισμός ε, του ΟΝΤΑΚ για το σκουμπρί δεν είναι καθόλου σκόπιμο και βεβαίως ε, αντίκειται σε κάθε πνεύμα συνεργασίας που είναι η βάση για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια ανεύθυνη συμπεριφορά μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για το απόθεμα στο άμεσο μέλλον. Εάν χρησιμοποιηθούν αυτά τα, αυτά τα ποσοστά από την Ισλανδία, θα ξεπεράσουν ε, και το, τις συστάσεις ε, το αλίας το, του 35% που έχει θέσει η ΆΙΣΕΣ. Οπότε θα υπάρξει απειλή για το απόθεμα. Οπότε νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά της Ισλανδίας ε, θα πρέπει να αναφερθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων προσχώρησης. Έχετε υπόψη ότι εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε διαδικασίες επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση ανεύθυνης ε, συμπεριφορά ή διαχείριση ε, των ε, αποθεμάτων. Είναι ώρα πια η Ισλανδία να κατανοήσει ότι όλα τα κράτη και τα κράτη-μέλη αλλά και οι υποψήφιες χώρες έχουν τους ίδιους κανόνες που πρέπει να σέβονται. Τώρα πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ μα και πρέπει να δείξουν καλή πίστη και την θέλησή τους να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Για τους ε, σοσιαλιστές, ο κύριος Τόμας. μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, οι προσπάθειε των Ευρωπαίων ε, ψαράδων για, τον, ε, για το σκουμπρί τα τελευταία χρόνια είναι υποδειγματικέ. Από το 2006 διαπιστώσαμε λοιπόν ότι επανέρχονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ε, τα αποθέματα σκουμπίου. Δυστυχώ δεν κερδίζουν αυτοί που έκαναν τις προσπάθειες. Διότι μόλις άρχισε να ανεβαίνει ο αριθμός των, των ε, ψαριών σκουμπριού, είδαμε ότι υπήρξε επίθεση από άλλες χώρες. Οι οικονομικές επιπτώσεις και η μείωση των ποσοστών για την Ευρώπη ήρθαν κατόπιν. Η οικονομική κατάσταση των αλλιών της Ένωσης βρίσκεται σε κίνδυνο σήμερα. Ολόκληρος ο, κλάδος, ο πελαγικός κλάδος της Ένωσης εμπλέκεται. Πάνω από 1500 σκάφη στη Γαλλία μόνο ψαρεύουν ε, σκουμπρί, κυρίως στα ανοιχτά της Βρετανίας. Μεταξύ αυτών πολλοί ε, εραστέχνες αλληλείς με αρνητικές επιπτώσεις και άμεσες μειώσεις ε, στις εκφορτώσεις. Αν η Ισλανδία και τα νησιά Φέρο αγνοούν την κατάσταση της βιομάζας, οι αλληλείς της Ένωσης θα γίνουν η μεταβλητή προσαρμογή της μείωσης του μέγιστου, της, της μέγιστης ποσότητας που είναι οι μόνοι που τηρούν. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε ένα κοινοθέντα, πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, η Ένωση πρέπει να λειτουργήσει ως ρυθμιστής και να υιοθετήσει κυρώσεις κατά των παρεκκλήσεων. Θα μπορούσαμε τα κράτη αυτά να τα εντάξουμε στα κράτη αυτών, μεταξύ των κρατών που δεν τη βιώσιμη αλληλεία. Δεύτερον, έχουμε συμφωνίες αλληλείας σε προνομιούχο καθεστώς με τις δύο χώρες αυτές, θα μπορούσαμε να τις αμφισβητήσουμε συνολικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ για τους πράσινους. Ο κύριος Χάτον, ένα λεπτό. Είναι δυσάρεστο να συζητούμε το ίδιο θέμα ξανά και ξανά χωρίς πρόοδο. Τουλάχιστον για το σκουμπρί ένα πολύ σημαντικό αλλιεύμα για τη σκοτία. Η Επιτροπή δεν μπορεί, παρότι λατρεύει τους κανονισμούς, δεν μπορεί να, να, να ρυθμίσει από ό,τι φαίνεται της, ε, την αλληλεία εξωτερικών δραστηριοτήτων. Η δύναμη που έχει η Κομισιόν εντός της Ένωσης δεν επηρεάζει από ό,τι φαίνεται καθόλου όταν προσπαθούμε να λύσουμε μια διεθνή διαφορά. Ο Υπουργός Αλίας της Σκοτίας πρότεινε να χρησιμοποιηθεί ένας διεθνής διαμεσολαβητής ενδεχομένω για να επιτευχθεί συμφωνία σε αυτό το δύσκολο ζήτημα. Λύνοντας με αντικειμενικό και ουδέτερο τρόπο το θέμα. Ελπίζω να μην εγκαταλείφθηκε αυτή η ιδέα γιατί ε, άκουσα μόνο άλλα εργαλεία που μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκαν. Ε, για τους συντηρητικούς, ο κύριος Γκέρλινγκ, 1,5 λεπτό η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε στον Ηνωμένο Βασίλειο όλα και σε άλλα κρατή μέλη με βέβαιη. Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο θέλουν να αγοράζουν και να καταναλώνουν ψάρια ε, τα οποία λέγονται από βιώσιμα αποθέματα και βασίζονται σε συστήματα πιστοποίηση για την επιλογή τους αυτή. Ο πολύ θρεπτικός, ε, ε, το πολύ θρεπτικό σκουμπρί άρχιζε να ε, εμφανίζεται πολύ συχνά σε διάφορα μενού, ήταν πιστοποιημένο, αλλά μετά από τη μονομερή δράση της ε, Ισλανδίας και των ίσων Φερόε ε, τα πράγματα αλλάζουν. Ενώ είναι πιο σκληροί οι κανόνε που πρέπει να ε, εφαρμόζει το Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπουμε να γίνονται αυτέ οι μονομερείς δράσεις. Ε, δεν βλέπουμε ότι θα υπάρξει άμεσα κατάρρευση του αποθέματο, αλλά στο μέλλον θα συμβεί αυτό. Αυτό που ήδη καταραίουν όμω είναι οι τιμέ. Οι Ευρωπαίοι αλήσει, οι οποίοι συμπεριφέρονται σωστά, σέβονται του κανόνε, παίρνουν τα μισά έσοδα από αυτά που είχαν πριν από δύο χρόνια. Όπω και οι συνάδελφοί μου ζητώ και εγώ λοιπόν και να μα απαντήσετε στα προφανή. Γιατί δεν εξασφαλίσατε μια βιώσιμη συμφωνία με Ισλανδία και Φερόε, απουσία της συμφωνίας αυτής. Πότε θα χρησιμοποιήσει η Κομισιόν της, ε, την εξουσία από ε, τις εντολές που πριν έξι μήνες σας έδωσε το Κοινοβούλιο για να λάβετε δράση. Έξι μήνες πριν, όχι έξι χρόνια πριν. Πρέπει να αλλάξουν οι συμπεριφορές αυτές. Πώς θα το επιβάλλετε αυτό και τι βήματα, τι μέτρα λαμβάνετε για να αναζωογονήσετε, για να αναβιώσετε τη Συμφωνία των Παράκτων Κρατών. Ευχαριστώ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 στενή συνεργασία μεταξύ όλων των ε, παράκτιων κρατών, ε, των λευτικών κρατών. Και αυτά γίνονται και ε, σε ό,τι αφορά την ρέγγα Ατλαντικού Σκανδιναβίας και μετά το 2010 όπως εξήγησε πολύ ξεκάθαρο ο κύριος Γκάλαχερ και για το σκουμπρί. Όμως ε, από το 2006 και μετά βλέπουμε να έχουν ε, αυξήσει από τα 4,5 περίπου στο 23% το μερίδιο του συμφερέως και από το 1 στο 23 Ισλανδία. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά ε, πλήττουν τη βιωσιμότητα των πόρων, των αλληλευτικών. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι τρόποι αλληλεία, δεν λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα άλλων χωρών, ούτε και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλη ε, δυσαρέσκεια και δυσφορία στον αλληλευτικό τομέα και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πρώτα απ' όλα για να υπάρχει αυτή η κουλτούρα ε, συμμόρφωσης προς τους κανόνες και από την άλλη πλευρά ε, σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές ποσοστώσεις και τα μέτρα διαχείρισης ξέρουμε ότι όλα αυτά θα τεθούν από αμφισβήτηση τελικά όπως και η ίδια αξιοπιστία ε, των μέτρων ελέγχου τα οποία υλοποιούνται. Πρέπει λοιπόν να ξαναβάλουμε, ε, να ξαναθέσουμε σωστά τους κανόνες του παιχνιδιού και περιμένω και η Επίτροπος να δείξει την απαραίτητη βούληση να βρούμε λύσεις. Ε, σωστά έχετε επιλέξει την οδό του διαλόγου, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη σας επίσης ότι είναι ανάγκη σε περίπτωση που δεν ευημερίσει ο διάλογος να αναλάβετε μέτρα και να βάλετε και προθεσμίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Καντέκ, 1,5 λεπτό. Επίτροπε, πρόεδρε, συνάδελφοι. Είμαι πολύ απογοητευμένος από το θέμα αυτό της κατανομής των ποσοστώσεων σκουμπριού. Η σύγκρουση μεταξύ Ένωσης Ισλανδίας ε, Φερόε αμφισβητεί μια μακρά συμφωνία διαχείριση των πόρων. Αυτή η μονομερή και ανεύθυνη αύξηση των ποσοστώσεων από τη Σφορέο και την Ισλανδία οδηγεί σε μια μη βιώσιμη εκμετάλλευση του σκουμπρού στην περιοχή. Η η αλληλεία έχει αυξηθεί το βαθμό που δεν είναι πλέον ε, βιώσιμη. Η Ισλανδία από πολλαπλασίες από 6-23 φορές την ε, αλληλεία. Πρέπει να προστατεύσουμε τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και πρέπει να, ξαναγεί, να ξαναρχίσει ο διάλογος γιατί διακυβεύεται το μέλλον των ωκεανών μας πρέπει στην Ένωση, στην Ένωση σεβόμαστε ποσοστώσεις και κανόνες. Τι κάνει όταν πρόκειται για αποθέματα που μοιραζόμαστε με άλλες χώρες. Ο κανονισμός του 2012 για τη μη βιώσιμη αλληλή επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων και την υλοποίηση μέτρων διαχείρισης ε, μη βιώσιμων μορφών αλληλίας. Τι περιμένει η Επιτροπή για να ξεκινήσει κυρώσεις που θα επέτρεπε ίσως να γυρίσουν, να ξανασκεφτούν τη λογική οι Ισλανδιακοί Φερόες. Η προκλητική αυτή στάση της Ισλανδίας μάλιστα έρχεται τη στιγμή που θέλει και περιμένει να γίνει μέλος της Ένωσης. Ευχαριστώ. Το Κάτσι Κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση που ζητούμε σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Οι μονομερείς αποφάσεις ε, της Ισλανδίας και των ε, νήσων Φερό για τις αλληλευτικές ποσοστώσεις ό,τι αφορά το σκουμπρί θα επηρεάσουν πάρα πολύ αρνητικά ε, και την οικονομία και το περιβάλλον των χωρών που αλλιεύουν το είδος αυτό. Η κατάσταση επιδεινώνεται. Οι μονομερείς αποφάσεις πλέον γίνονται κοινή πρακτική. Έχουμε ανεύθυνο υπολογισμό και καθορισμό ποσοστώσεων. Θα πρέπει να γίνει πιο ε, δίκαιη κατανομή και θα πρέπει να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στις αντιδράσεις μας. Έχουμε ε, επανειλημμένες παραβιάσεις. Δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε τον ενδεχόμενο της επιβολής κυρώσεων. Η Κομισιόν ε, είναι πάρα πολύ σοβαρή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και είμαστε πρωταθλητές στην οικολογική αλία, στη βιωσιμότητα ε, γιατί έχει μεγάλη ευαισθησία η Κομισιόν, αλλά δεν κάνει κάτι για τους ε, εκτός. Τι κάνετε στην προκειμένη περίπτωση, τι αποτελέσματα έχετε επιτύχει. Δεν πρέπει να υπάρξουν και κάποια κίνητρα που θα πρέπει να δώσουμε σε αυτές τις χώρες συζήτηση που θα έχουμε μαζί τους. Ο κ. Νικολέσκου τώρα. Μη Κολέσκου. Ε, Καλωσορίζω τις θέσεις του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και συμφωνώ με τους συναδέλφους που υπογράμμισαν την ανάγκη να έχει μια σταθερή αποφασιστική θέση η Ένωση. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι μοναδική. Χρειαζόμαστε την ίδια στέρεη και αποφασιστική στάση της Ένωσης στην αλληλεία στον εύξηνο πόντο όπου η αλληλευτική ε, δραστηριότητα είναι πολύ περίπλοκη γιατί μόνο δύο από τα έξι παράκτια κράτη είναι μέλη της Ένωσης. Πρέπει να είμαστε πολύ δραστηριοί εκεί. Δυστυχώς ωστόσο ο διάλογος με τις τρίτες αυτές χώρες παράκτιες του εύξηνου πόντου δεν είναι ικανοποιητικός. Κλείνοντας να σας πω ότι η Κίνα ψαρεύει 12 φορές περισσότερα ψάρια από όλα τα άλλα κράτη της, ε, των Ηνωμένων Εθνών. Τα περισσότερα προέρχονται από την Αφρική αλλά αυτό δεν είναι παρηγορητικό. Χρειαζόμαστε εταίρους που θα κάνουν θυσίες στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Πρόσφατα κάναμε μια συζήτηση για τη νέα ληφτική πολιτική που πρέπει να είναι βιώσιμη, αλλά έπρεπε να διατηρεί και το εισόδημα των αλλιέων. Τα πράγματα όμως έχουν ε, ε, ξεφύγει πια ε, με τούτε δύο χώρες, ε, την Ισλανδία και τις νήσους Φερόε. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό που κάνουν στις κατοχώρες. Οι τιμές πέφτουν με βάση αυτά που έχουν κάνει. Οπότε ρωτώ, πού έχουμε φτάσει με τα βήματα που έχετε κάνει εσείς, πόση πρόοδο έχετε επιτύχει και επίσης όταν έχουμε μια κοινότητα αξιών, μια συμφωνία είναι συμφωνία. ισχύει και για τη συμφωνία και για την Ισλανδία, είτε αυτή είναι προσχωρή είτε είναι κράτος μέλος. Και δεν μπορεί η Ισλανδία να συνεχίζει μονομερό να δρά, πρέπει να το καταλάβει. Στήλερ. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριο ε, Φανίστερ Ρόι. Η Κομισιόν θα σκεφτεί την ε, πρόταση του κύριου Χάριστον για έναν διεθνή διαμεσολαβητή. Νομίζω ότι αυτό είναι μία από τι ανησυχίε ε, που είναι αρκετά σκόπιμο να τι σκεφτούμε. Και επίση, όπω είπαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, οι τρέχουσε διαπραγματεύσει με την Ισλανδία και την προσχώρηση τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζονται. Και όπω ξέρετε, κύριε Επίτροπε, οι Ισλανδικέ εκλογέ είναι την επόμενη εβδομάδα. Θεωρείτε ότι μόλι γίνουν οι εκλογέ θα υπάρξει ίσως ευκαιρία για περισσότερη πρόοδο σε τούτο το θέμα. Η Ισλανδία ε, ακόμη δεν έχει ασχοληθεί με, την, ε, με το θέμα της αίτησή τη ε, για την ε, αλληλεία. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι επίγον και πρέπει να το δούμε. Το έχουν πει πολλοί συνάδελφοι. Είναι τελείως μη βιώσιμο αυτό που έκανε και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει δράση απέναντι σε αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Davis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Στάιλερ όντω έκανε ένα, είπε κάτι πολύ σωστό. Είναι γνωστή η Ισλανδία. Ε, προσπαθεί βιώσιμα να αλλιεύσει, αλλά η φήμη τη θα καταστραφεί με βάση αυτό το θέμα του, με το σκουμπρί. Καλωσορίζω λοιπόν ε, την ε, προσχώρηση τη Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ξέρουμε ότι οι διαπραγματεύσει ακόμα τρέχουν και είναι και ευαίσθητε. Έχουν και τι εκλογέ. Βεβαίω, δεν είμαι εγώ αυτό που, θα ζητήσω από την Επίτροπο να μου πει αν την πιέζουν ε, με κάποιο τρόπο, αλλά συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Στήλερ. Κυρία Επίτροπε, θεωρείτε ότι αν δεν είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τι διαπραγματεύσει για να εξασφαλίσουμε βιώσιμη συμφωνία αλληλία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισλανδία. υπάρχει κίνδυνο να καταρρεύσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Εντάξει, δεν θα, δεν σας πιέσω, δεν θα, ρωτήσω αυτό που θέλω, δεν θα το πιέσω. Ευχαριστώ. Η Επίτροπος κ. Δαμανάκη έχει Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να παρέμβει στη προεκλογική εξαρτία της Ιλλανδίας και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω ευθύς εξ αρχής όμως τώρα να εστιάσω στο θέμα που μας απασχολεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρεμβάσεις σας. Θέλω να επαναλάβω ότι κάνουμε πολλά για να ασκήσουμε πιέσεις ε, στην Ισλανδία και στα νησιά Φερό για να ξανακαθίσουν ε, στο τραπέζι και να υπάρξει συμφωνία και για τα δύο αποθέματα, δηλαδή του Σκουμπρί και τη ε, Ρέγκα Ατλαντικού Σκανδιναβία. Προσπαθούμε και για τα δύο αποθέματα. Με τι μέσα, με τι τρόπου. Πρώτον, με το διάλογο, διμερείς επαφές, ε, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το ζήτημα αυτό και σε, να το θέσουμε και σε διεθνή βήματα συζήτησης όποτε και όπου μπορούμε. Δεν αποκλείουμε οποιαδήποτε πρόταση. Έχουμε λάβει την πρόταση για τον ενδεχόμενο ορισμό μεσολαβητή, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν επιλέξουμε την οδό αυτή, όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι τελικά θα δεχθούμε και το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πιστούν όλοι για να συμφωνήσουν. Δεν θα είναι εύκολο λοιπόν. Δεν το αποκλείουμε όμως, όπως και δεν αποκλείουμε τίποτε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα για όλους εσάς, σχεδόν όλους, για να μην πω όλοι οι ομιλητές τουλάχιστον υπογράμμισαν την ανάγκη να εφαρμοστεί αυτό ο νέος κανονισμός για τις εμπορικές κυρώσεις. Το μήνυμα ελήφθη, αλλά θέλω να επαναλάβω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια συγκεκριμένη νομική βάση έχοντας υπόψη μας και το χρονοδιάγραμμα. Και επίσης χρειαζόμαστε συμμάχους. Εξού και ε, όταν μιλούσα για το σκουμπρί σας είπα ότι θα το συζητήσω ξανά το θέμα με τον Νορβηγό Υπουργό την επόμενη εβδομάδα. Την Νορβηγική Υπουργό θα συναντήσω Τετάρτη συγκεκριμένα και μετά θα σας ενημερώσω για την απόφαση που θα ε, λάβουν. Γιατί θα πρέπει να έχουμε στο πλευρό μας και τους Νορβηγούς, τους χρειαζόμαστε. Αλλιώς το αποτέλεσμα δεν θα είναι τόσο καλό όσο θα θέλαμε. Τώρα, για την άλλη υπόθεση, δηλαδή την Ρέγκα, Ατλαντικού Σκανδιναβία, σας είπα πολύ ξεκάθαρα ότι νομίζουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο. Εγώ έχω δώσει το πράσινο φως να ο εσωτερικά η διαδικασία στη, στο επίπεδο της Κομισιόν για την υλοποίηση του εμπορικού μέσου, δηλαδή για την επιβολή εμπορικών κυρώσεων στα νησιά Φερόε, για την προκειμένη περίπτωση, επειδή εγκατέλειψαν ε, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Ολοκληρώνει τη συζήτηση και προχωρούμε το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης έκθεση Τσίστερ για την Ευρωπαϊκή